Αγαπητοί συνάδελφοι, ήγηκε η ώρα. Σα καλώ να καθίσετε για να αρχίσει η συνεδρίαση. La séance est ouverte. Je vous prie de Άρχεται η συνεδρίαση. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι χάνω σιγά σιγά τη φωνή μου. Στα γαλλικά λέμε κατά λέξη ότι αισθάνομαι σαν να έχω μια γάτα στο λαιμό. Και στην Αγγλία τι λέμε, ένα βάτραχο στο λαιμό, a frog in the throat. Έκτακτη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών, όπου θα ασχοληθούμε με πολλές και σημαντικέ ψηφοφορίες. Ας διασφαλίσουμε καταρχάς ότι συμφωνείτε με την, με την διάταξη ως έχει. Συμφωνείτε από ό,τι φαίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Θα ήθελα να αφαιρθώ στον πρώτο δημοσιονομικό τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα την 5η, 27 Μαρτίου, παρουσία του Επιτρόπου Ότιγκερ, της ε, Μαλτέζικης Προεδρίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών Εντουάρ Σίκουνα και παρουσιάστηκαν οι κατευθύνες γραμμές που είχε εγκρίνει το Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη δική της την πλευρά παρουσίασε τις δικές της κατευθύνες γραμμές που εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της 15ης Μαρτίου. Μια κοινή δήλωση ακολούθησε στη συνέχεια με το χρονοδιάγραμμα Τη δημοσιονομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί εγκρίθηκε και αυτό το χρονοβιογράμμα και σας κοινοποιήθηκε. Τέλος, κάναμε μία αποτίμηση της κατάστασης όσον αφορά του εκρεμεί διορθωτικού προπολογισμού και του μελλοντικού διορθωτικούς προπολογισμού και όσον αφορά τι χρηματοοικονομικές επιπτώσει για τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένω ο Ζίκρφιτ Μούρεσαν θέλει να πάρει το λόγο, ο οποίο είναι ο γενικός ηγητή μα όπως ξέρετε, για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα. Έχουμε τον νεαρινό τριμερή διάλογο με την Προεδρία και τον Επίτροπο Έτιγκερ και εκεί είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του επομένου έτους με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο στην Ολομέλεια βασικές μας προτεραιότητες ανάπτυξη και δουλειές και δύο ασφάλεια των πολιτών και επαναλάβαμε το ότι θα πρέπει να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση για έρευνα, καινοτομία, υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεργία των νέων. Ε, πολύ σημαντική η προτεραιότητα του Κοινοβουλίου. Επίσης είπαμε ότι περιμέναμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να είναι έτοιμη να βοηθήσει τους αγρότες αν προκύψει κάποια κρίση και για το θέμα της ασφάλειας επαναλάβαμε την στήριξή μας για την προπαρασκευαστική δράση για την άμυνα και για την ενίσχυση της νότιας και ανατολικής άμεσης γειτονίας της Ένωσης για να υπάρχει καλύτερη προστασία των συνόρων και περισσότερη ασφάλεια για τους πολίτες της Ευρώπης. Η Κομισιόν σκοπεύει να υποβάλει ένα σχέδιο προπολογισμού πριν από το τέλος Μαΐου και το χρονοδιάγραμμα που ανέφερε ο Πρόεδρος που εγκρίναμε για την διαδικασία του προπολογισμού είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρότειναν οι συντονιστές κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε την θέση μας στην δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου η διαβούλευση θα ξεκινήσει 31 Οκτωβρίου και θα τελειώσει 20 Νοεμβρίου. Πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι θα έχουμε δύο συναντήσεις για τη συνδιαλλαγή. Πρώτη στις 9 Νοεμβρίου και η δεύτερη, είναι σημαντικό αυτό, 17 Νοεμβρίου, Παρασκευή. Αμέσως μετά το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες. Να ξέρουν λοιπόν οι βουλευτές ότι θα έχουμε αυτή ακριβώς συνεδρίαση αμέσως μετά την εβδομάδα του Στρασβούργου. Αυτά από μένα κύριε Πρόεδρε. Merci, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Εισηγητή. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Μπορούμε όμως ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Σας κάνουμε μια δοκιμή με τις κάρτες σας προκειμένου να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Α κάνουμε λοιπόν μια δοκιμή. Χρησιμοποιήστε τι κάρτε σα. Άρτε ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Όχι. Ναι. Πολύ ωραία. Πέρας. Εσείς δεν έχετε κάρτα, η κυρία Πιτσέρνο. Επομένω θα ψηφίσετε διανατάσεως. Και εσείς, πολύ ωραία, λοιπόν θα προσέχω και τους δυο σας να δω πώς ψηφίζετε. Και προφανώς θα προσθέτω κάθε φορά τις δικές σας ψήφους στο τελικό αποτέλεσμα. Ο Ρίτσαρτ Άσουορθ ε, έκανε κάθε το δυνατό για να έρθει σήμερα, αλλά αντιμετώπισε κάποια προβλήματα με την πτήση του, η οποία καθυστέρησε λόγω των ατμοσφαιρικών συνθήκων, της έντονης ομίχλης και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να φτάσει στο Στρασβούργο πριν από τις 11 το βράδυ σήμερα. Αν αναβάλαμε την ψηφοφορία για αύριο το πρωί, θα είχε περιπλέξει πολύ περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά το πέρασμα της έκθεσης αυτής στην Ολομέλεια. Με τη δική του την άδεια λοιπόν, την άδεια του κυρίου Άσπορθ μπορούμε να προχωρήσουμε σήμερα στην ψηφοφορία για την έκθεση αυτή προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 και να ψηφίσουμε για το αποτέλεσμα της διαλλαγής της 5ης 28 Μαρτίου 2017 0 3% η αύξηση προβλέπεται εδώ πέρα. Ο κύριος Λούκε αντικαθιστά τον κύριο Άσχορθ και θα ψηφίσει εξ ονοματός του. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε καταρχάς για την συμφωνία αυτή καθεαυτήν με το παράρτημα υπαριθμών 1 όπου προβλέπονται συγκεκριμένε τροποποίησεις. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, της πρότασης αυτής διανατάσεως. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές το παράρτημα περιθμών 1 εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες του εισηγητή, παράρτημα περιθμών 2 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές και το παράρτημα 2 εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις υπόλοιπες τροπολογίες. Ορισμένες, όπως βλέπετε, καλύπτονται από τη συμφωνία την οποία μόλις τώρα εγκρίναμε. Τροπολογία 10, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται 11 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 20 κατά. Τροπολογία υπέρ 11 υπέρ Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Οι 13 και 14 καλύπτονται από την προηγούμενη ψηφοφορία μας. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Στον αφορά τροπολογία 17, λέει ο Πρόεδρος, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ. το όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση γεντροπολογή 24, άρτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ και 11 κατά. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 27. Η 24 όμως εγκρίθηκε, λέει ο πρόεδρος. Επομένω η τροπολογία 27 καταπίπτει και περνάμε στην τροπολογία 28 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 τώρα όπου έχουμε ψηφορία σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ μάλλον καταπίπτει 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 37 με προφορική τροπολογία του κυρίου Νεγκρέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, μάλλον καταπίπτει, γιατί εγκρίθηκε 37. Περνάμε σε 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβαστική τροπολογία παριθμών 1, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ και 12 κατά. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 έναντι 14. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 55 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 κατά 14 υπέρ. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 64 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 66 με τεχνική προσαρμογή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 67 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 67 πάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, άρθρη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 17 κατά, 73 υπέρ, κατά. Στο συγγνώμη 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 74 καταπίπτει. Οι 75 και 76 τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά στο παληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία 77 πέρας απορρίπτεται 18 προς 15 78 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται η 79 υπέρ. Να το επαληθεύσουμε. Πολύ ωραία. Για την 78 λοιπόν, άρτε ψηφοφορία. Απορρίπτεται 18 προς 13. Η 79 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 84 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. 85 τώρα υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, την ψηφίζουμε κανονικά. Η 83 εγκρίθηκε, να έχετε δίκιο, σας το συγγνώμη. Επομένως η τροπολογία 85 καταπίπτει, 86 και 87 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ μάλλον καταπίπτει υπέρ μάλλον για το 89 υπέρ υπέρ της 89 παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία παριθμών 3, άρχιτη ψηφοφορία. εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 2 εποχές. Προπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Να σηκώνετε καλά το χέρι σας παρακαλώ πολύ. 101. Καταπίπτει. ήταν συμβατή με την 99 για την 101 υπέρ κατά εγκρίνεται 104 τώρα σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 105 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται 111, 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Βασική τροπολογία 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 119 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 112 λέει ο πρόεδρος συγγνώμη 122 διορθώνει τροπολογία 122 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ε, να το επαληθεύσουμε πρώτο τμήμα της 122 ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21 προς 14. Δεύτερο τμήμα της 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 146 σε τρία τμήματα το συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρτη ψηφοφορία εγκρίνεται 27 ψήφοι υπέρ και 9 κατά ψηφίσαμε την 134 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος. 136 και 137 τώρα ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. 136-137 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνονται με 26 ψήφους υπέρ και 9 κατά. 138 μάλλον έχει καταπέσει. 139 λοιπόν και αυτή έχει καταπέσει. Η 140 καταπίπτει και αυτή, η 141 καταπίπτει και αυτή, 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 144 τώρα υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε την 144. Πέρας. Εγκρίνεται. Να σηκώνετε καλά το χέρι σας παρακαλώ πολύ. 145 υπέρ. Μάλλον έχει καταπέσει. Σας το συγγνώμη ο πρόεδρος. Στην 146 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 147 σε δύο τμήματα. Θέλετε να επαληθεύσουμε το τρίτο τμήμα της 146. Πολύ ωραία. Άρθε ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 17 κατά. Η 147 τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Δεν σηκώστε πολύ το χέρι σας. Πρώτο τμήμα της 147 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 σε δύο τμήμα, τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 149 άρτη ψηφοφορία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 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά εγκρίνεται 161 υπέρ μάλλον καταπίπτει 162 καταπίπτει και αυτή και περνάμε έτσι στη συμβαστική τροπολογία περιθμών 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά στο επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά ψηφοφορία για την 173 πέρας σας το συγγνώμη εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ και 10 κατά 174 υπέρ κατά αποχές είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 174. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ και 10 κατά. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176 και 177 μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 178 καταπίπτει. Η 179 καταπίπτει επίσης. Το ίδιο και 180 και 181 και 182 έχει αποσυρθεί. 183 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 185 τώρα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 186 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187 και 188 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτονται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 192 και 193 από κοινού έχουν τον ίδιο στόχο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 194 μάλλον καταπίπτει. Η 195 καταπίπτει επίση. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 203 υπέρ. Συγγνώμη, καταπίπτει 203 και 204. Περνάμε τώρα στις λογικές σκέψεις 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 4 άρτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ και 16 κατά τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά εγκρίνεται το σύνολο τώρα της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε Ψηφίζουμε μονομαστική κλίση, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ και 4 κατά και 2 αποχές. Ας συγχαρούμε τον εισηγητή μας και τους κοιόδης εισηγητές. για την έκθεση του Χωσέ Μανουέλ σε σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν υπάρχουν τροπολογίες. Με ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Εκθέση Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Κύπρο και την Πορτογαλία. Πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια. Τώρα του κυρίου, η έκθεση του κ. Γκάγερ, γενικός, γενικού εισηγητή, διορθωτικός προϋπολογισμός νούμερο 1. Υπάρχει μια τεχνική τροποποίηση, δεν θα γίνει ψηφοφορία. Μάλλον γίνεται μόνο ονομαστική σε όλο το κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 35 υπέρ, μια κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Για την έκθεση του ε, Βίκτορ Νεγκρέσκου, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, έχουμε τέσσερις τροπολογίες. Τροπολογία 1 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου, ονομαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 30 υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Για την έκθεση του Σίγφριτ ε, Μουρεσάν, μακροοικονομική αρρωγή για την ε, Δημοκρατία της Μολδαβίας, τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την τροπολογία 6 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ε, ε, ψήφους κατά, 17 ε, υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 Καταπίπτει 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω την πλειοψηφία, οπότε θα κάνουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Για το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε νομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ κατά 6. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκθεση της κυρίας Νιριάντα προώθηση του διαδικτύου στις τοπικές κοινωνίες. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε. Την 42. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 19 κατά και 15 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 8. Προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για τις αιτιολογικές σκέψεις, η τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 σταματάει η ψηφοφορία γιατί καλύπτεται αν εκκριθεί η 7. Τροπολογία 2, συμβαστική, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβαστική 3. Όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 17. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε επειδή είναι συμβαστική. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 28 κατά, 8 υπέρ. Ωραία. Τροπολογία 2. Υπέρ. Τη 2. Ναι. Γιατί ήταν στη συμβαστική 5, αφού δεν ψηφίσαμε την 5, πρέπει να ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες που κάλυπτε. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Α, απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 3. Προφορική. Υπέρ. Κατά. Και ποιος από... Εγκρίνεται. ...30 και 31 καταπίπτουν... ...συμβαστική 6... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...συμβαστική 7... ...υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλύπτει και την τροπολογία 13 που αφήσαμε πριν για μετά όπως και την 11 και την 37 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 11 έχει καλυφθεί. Στο σύνολο του κειμένου ψηφίζουμε τώρα, όπως τροποποιήθηκε, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. τμήμα 3 του Γενικού Προϋπολογισμού μας ε, προτείνουν μεταφορά για το ε, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μεταφορά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Για τα άλλα τμήματα του κυρίου Ταράν δεν υπάρχει αίτημα μεταφοράς, ούτε αίτηση για πίστοση για τα έπιπλα. Τελειώσαμε. Για τα ακίνητα. Ε, τελειώσαμε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα στη συνεδρία σας. Καλό βράδυ.